και όλο πιο δύσκολες στην Ουκρανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως στην μεγάλη του πλειοψηφία επιμένει για την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία στην Ουκρανία. Σε πολλά ψηφίσματά μας έχουμε ήδη πει ποια είναι η απόψή μας. Εξάλλου θα το συζητήσουμε και αυτή τη βδομάδα, ότι δεν θεωρούμε νόμιμη την εισβολή αυτή στην Κρυμαία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια στρατηγική που θέλει να κόψει τη χώρα σε κομμάτια. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές του διεθνούς δικαίου και πρέπει να αποσυρθούν τα στρατεύματα από τα εδάφη της Ουκρανίας. Πρέπει να αποφύγουμε κάθε αποσταθεροποίηση της χώρας. Είμαστε όλοι εδώ βέβαιοι, σίγουροι για την ευθύνη που έχουμε. Είμαστε υπέρ κάθε δραστηριότητας που έχει σαν στόχο να στηρίξει την κυβέρνηση της Ουκρανίας για να υποστηρίξει την ακεραιότητα της χώρας, να στηρίξει τα σύνορά της και να μπορέσει να υπάρχει διάλογο στο εσωτερικό της χώρας. Θέλουμε η Ουκρανική οικονομία επίσης να σταθεροποιηθεί. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά τα κοινωνικά προβλήματα στη χώρα αυτή. Και γι' αυτό ακριβώς είμαι ευτυχής για την απόφαση που πήρε το Συμβούλιο σήμερα για να δοθεί ένα δισεκατομμύριο βοήθεια στην Ουκρανία όπως είχαμε ήδη συζητήσει εδώ την προηγούμενη φορά. Πρέπει πραγματικά να δράσουμε μαζί. Θα εγκρίνουμε ψήφισμα την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Θέλει επίσης να στείλει και μία αντιπροσωπεία στις εκλογές που θα γίνουν το Μάιο στη χώρα. Εκλογές οι οποίες πρέπει να γίνουν με δίκαιο τρόπο, ελεύθερα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι οι εκλογές αυτές θα οδηγήσουν σε ένα κεφάλαιο ελευθερίας και ειρήνης στην ιστορία της Ουκρανίας για να μπορέσει η χώρα αυτή να ζήσει εν δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, 6 με 7 Απριλίου τη νύχτα αυτή έγιναν οι συζητήσεις για την γενοκτονία στη Ρουάντα. Η επέτειος αυτή πρέπει να μας υπενθυμίσει ότι μέσα σε μια περίοδο 100 ημερών πάνω από 8.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σκοτώθηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οι γυναίκες και παιδιά. Μωρά, μάλιστα. Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν, σκοτώθηκαν από τους γειτονές τους ή από αυτούς που υποτίθεται ότι ήταν οι φίλοι τους. Και αυτό απλώς και μόνο επειδή ανήκαν σε μια διαφορετική εθνική ομάδα. Η διεθνής κοινότητα τότε έστρεψε το βλέμμα αλλού. Δεν στάθηκε στο ύψος των ευθυνών της τότε. Η γενοκτονία αυτή προβλέφθηκε από ανθρώπους και μπορεί να επαναληφθεί ανα πάσα στιγμή. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Χθε ήταν η Ρουάντα, η Σρεμπρενίτσα. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει την επόμενη φορά κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει ένα μάθημα από αυτή τη γενοκτονία στη Ρουάντα είναι αυτό το μάθημα. Ότι δεν μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα αλλού. Και έτσι σε σχέση με την ανάμειξη στα εσωτερικά μιας χώρας δεν είναι ακριβώς αυτό. Και οι υπεύθυνοι για τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να προσάγονται στη δικαιοσύνη. Και αυτό αφορά και τον δικτάτορα, την δικτατορία στη Συρία δεν μπορούν να υπεκφύγουν της δικαιοσύνης. Γι' αυτό είναι τόσο πιο σημαντικό το εθνικό και το διεθνές δίκαιο να μπορεί να επιβληθεί. Και το διεθνές ποινικό δικαστήριο πρέπει περαιτέρω να ενδυναμωθεί βρήκαν οι κάτοικοι της Ρουάντα τον δρόμο τους και είναι δυνατόν να υπάρξει συμφιλίωση, το κατέδειξαν αυτό. Εξ ονόματος του Ευρωκοινοβουλίου θέλω να πω στους κατοίκους της Ρουάντα ότι θέλουμε να τους υποστηρίξουμε σε αυτή την πορεία τους για μια ειρηνική συμβίωση και πορεία της χώρας τους επεξεργάζεται αυτό το παρελθόν της ε, η Ρουάντα για να το ξεπεράσει και πρέπει πραγματικά οι εγκληματίες οι οποίοι έχουν ε, διαπράξει τέτοια εγκλήματα πρέπει να τιμωρηθούν και πρέπει να βοηθήσουμε επίσης μέσω οικονομικής σταθερότητας να μπορεί να βρει την εσωτερική ειρήνη η χώρα αυτή. Έχουμε την αλληλεγγύη που εκφράζουμε ως Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα θύματα και προς τους οικείους τους. Και κάτι θλιβερό όσον αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να σας ανακοινώσω την προηγούμενη Πέμπτη η η μετά από μακρά ασθένεια 66 ετών απεβίωσε. Το 2011 η Ντομινίκ ήταν από πλευρά της, του αξιώματος του συνήγορος του πολίτη και έδωσε αγώνα για τον, την ισότητα και ήταν και ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή και ε, ήταν και δημοσιογράφος και έγινε, ε, ακολούθησε το αξίωμα του πατέρα του ως δήμαρχος της ε, Τουλούζ. Σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία ήταν ε, ευρωβουλευτής και είχε μακρά θητεία. Πολύ θα τον θυμόσαστε ως ένα πολύ σεβαστό άτομο που ήταν πραγματικά γενναιόδωρος και είχε πάντα καλά λόγια να πει σε όλους. Ένας άνθρωπος ε, που ε, ήταν υπέρ του διαλόγου και ήταν ε, και υπεύθυνο για το Institut du Monde Arabe, το Ίδρυμα για τον Αραβικό Κόσμο. Πολύ δύσκολες καταστάσεις αντιμετώπισε και έπρεπε να υποστεί κατά τη διάρκεια του βίου του. Και επιθέσεις που υπέστη που αποδείχθηκαν ότι ήταν, ε, πραγματικά δεν ευσταθούσαν. Θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήριά μας προς τους οικείους του. Παρακαλώ <clears throat> για τα θύματα της Ρουάντα και το συνάδελφό μας να εγερθούμε και να αποτίσουμε τιμής για αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις για τη Δευτέρα Απριλίου δεν υπάρχουν. Για τα πρακτικά ή για κάτι άλλο. Τότε τα πρακτικά λοιπόν της ε, Δευτέρας Απριλίου εγκρίνονται. Για διαδικαστικό εσείς. Παρακαλώ. Για διαδικαστικό μάλιστα. Θα ήθελα να ζητήσω το εξή, Πρόεδρε. Στι 10 Απριλίου, πριν από τέσσερι ημέρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλε, είχαμε μια ακρόαση των ε, ε, πρωτοβουλειών των πολιτών. Ήταν μια πολύ επιτυχή πρωτοβουλία των πολιτών. Και ο πρόεδρο των Σοσιαδημοκρατών είχε αποστείλει και Διακόπτει ο Πρόεδρος. Με συγχωρείτε να σας διακόψω. Παρακαλώ πρώτα να καλύψουμε τα δικαιώματα.